must be the anti-Gazprom amendment. Abstimmung ist geschlossen. Es ist mit 23 zu 20 angenommen worden. 95. Yeah. 94 we cannot vote because two was also agreed. It was 95, now we come to 96. Who is in favor?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 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 37 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 38 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι έχει να δεκτεί 39 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 40 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 41 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 46 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 47 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 48 υπέρ κατά αποχές απερίφθη να επελθεύσουμε Μα το ΕΛΚ έχει αρνητικό πρόσημο εδώ. Το ΕΛΚ έχει αρνητικό πρόσημο. Σαράντα οχτώ υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. weiß ich das. Der Obergasplan. Da kann man schon vorstellen, was der Unterschied ist. Ja. Tja. Herr Berichterstatter, dann müssen Sie doch... Πρέπει να συνεννοηθείτε με τους συντονιστές σας, κύριε συντονιστά. Κύριε συντάκτα. Εγκρίνεται λοιπόν. 49. Υπέρ κατά αποχές απερίφθη 50 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 51 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 52 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 53 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 54 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά να με βοηθήσουν οι σοσιαλιστές παρακαλώ πρέπει να πάρω μια απόφαση μεταξύ δύο, δύο ΕΛΚ ε, επιλογών του ΕΛΚ λοιπόν παληθεύουμε ηλεκτρονικά την 56 Ήξερα ότι ο Σάριος Βόλος και συμφωνούσε στα θέματα του φυσικού αερίου με τους σοσιαλιστές. Πέρας. 15 υπέρ, 28 κατά, απερίφθη. 57 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 58 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. 59 υπέρ, κατά σε απερίφθη. Συμβαστική υπαριθμών 1. Αργά στον κατάλογο φτάνει, πάση περιπτώσει, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και πάμε στην 63 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 64 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη, 65 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη, αν μπλοκ της Ζαμβάσκη συμφωνείτε μέχρι το τέλος. Κυρία Λέζινγκ, σα ευχαριστώ πολύ για το πνεύμα συνεργασίας. 66 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 67 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 68 υπέρ κατά αποχέ. απερίφθη, 69 υπέρ κατά απόχε. απερίφθη, 70 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 71 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 72 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 73 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 74 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 75 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 76 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και κυρία Λούζιν εσείς τώρα ήσασταν κατά μόνο 78 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 79 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 80 ε, υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 81 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 82 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 83 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και 89 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές απερίφθη παριθμόν 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά 91 υπέρ κατά απερίφθη τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ αρχίτε πέρασε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 32 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται α, συγγνώμη 35 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 36 Στο κυρίου Επιτίδιο Until 45. Do you agree? Μέχρι την 45 να του ψηφίσουμε μαζί, συμφωνείτε? Από την 36 μέχρι την 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Φτάνουμε στην τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όταν ε, γράφει ότι είναι του εισηγητή, ε, έχει τρεις ψήφους παραπάνω η, η τροπολογία. 11 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Το δέχεστε. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14. Καταπίπτει. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φτάνουμε στην 5. Ευχαριστώ κύριε Πρέντα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά 17, τι είπα εγώ. Ε, κοντά έπεσα. Δεκαεπτά λοιπόν. Κατά. Αποχές. Ποιος είναι υπέρ. Απορρίπτεται. 18 ε, κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. It's closed. Λήξη της ψηφοφορίας. 23 ψήφοι υπέρ, 22 κατά. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Την 21 ελέγχουμε. I Λήξη της ψηφοφορίας. 16 υπέρ, 30 κατά. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. 23 υπέρ. Κατά. Μόλις ψηφίσαμε την 22. Μόλις ψηφίσαμε την 22. Η ηλεκτρονική επαλήθευση της 22. Uh, Ελέγχουμε το αποτέλεσμα της 22, διότι θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι καταλάβατε καλά. Περί τίνος πρόκειται. It's Λήξη της ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 22 κατά. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 26 καταπίπτει. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έναρξη της ψηφοφορίας. Die Abstimmung ist geschlossen. Λήξη της ψηφοφορίας. 39 39 ψήφοι υπέρ, 7 ψήφοι κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε συντάκτη. Wir kommen jetzt. Προχωράμε τώρα στην ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Χάν. για θέματα της αρμοδιότητάς του και ιδιαίτερα όσον αφορά την, ε, την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Δεν ε, θα σας διαβάσω όλες τις σημειώσεις που έχω μπροστά μου. Θα του δώσω κατευθείαν το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν σαφής η εντολή σας. Ούτε και εγώ θα αναφερθώ σε όλες ε, τις χώρες ε, μία προς μία. Επιτρέψτε μου όμως να πω λίγα λόγια για την Τουρκία. Η είπατε εκπρόσωπος ε, και εγώ βρεθήκαμε εκεί την προηγούμενη Παρασκευή. Μετά από όλες τις εντάσεις που υπήρξαν ανάμεσα στην Ευρώπη και την Τουρκία, Ε, είχαμε μια σχετικά αρμονική συνάντηση. Νομίζω ότι η κατάσταση γενικά και θα έχουμε την ευκαιρία να το συστήσουμε αυτό αύριο στην Ολομέλεια, είναι μάλλον ασαφής. Νομίζω ότι όλοι βρισκόμαστε σε κατάσταση σοκ οι συνάδελφοι στην Τουρκία ίσως ακόμα περισσότερο και από εμά. Αλλά η επίθεση αυτή στην ε, τουρκική δημοκρατία έχει καταδικαστεί ε, σε όλο τον κόσμο. Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι Έχουμε διαφορές με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι χώρα υποψήφια, γι' αυτό ε, αναμένουμε υψηλά πρότυπα από τη χώρα αυτήν. Και κατά την προετοιμασία της, ε, του πραξικοπήματος ε, και κατά την δίωξη των υπόπτων για συμμετοχή στο πραξικόπημα, Περιμένουμε διαφάνεια στη διαδικασία κατά τη δίωξή τους. Πριν ε, σχεδόν ε, δύο μήνες συνέβη αυτό και είχαμε συζητήσεις ε, με τον Υπουργό για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις και με τον Πρωθυπουργό και μας διαβεβαίωσαν ότι θα σεβαστούν ε, τα πρότυπα αυτά. Έχουμε ε, ανταλλαγές απόψεων με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο εξετάζει και παρακολουθεί προσεκτικά τα θέματα αυτά. Από ό,τι γνωρίζω, η Τουρκία δεν έχει απαντήσει στην ε, πρόταση που της έγινε σχετικά με παρακολούθηση της διαδικασίας. Σίγουρα θα είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση τις επόμενες μέρες και τις επόμενες εβδομάδες. και αρχές Νοεμβρίου θα ε, παρουσιάσουμε ε, την έκθεση προόδου, οπότε θα πρέπει να, να επικαιροποιηθούν ανάλογα τα σχετικά κεφάλαια. Ε, στα, πέρα από τα γεγονότα αυτά έχουμε στενή συνεργασία με την Τουρκία στο θέμα της μετανάστευσης, έχουμε τη συμφωνία για τους πρόσφυγες. Άσχετα από τα γεγονότα της 15ης-16ης ε, Ιουλίου, ε, τα πράγματα στον τομέα αυτών ε, εξελίσσονται ομαλά. Βλέπουμε εφαρμογή της συμφωνίας. Ο αριθμός των μεταναστών που φτάνουν από την Τουρκία στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, έχουν μειωθεί σημαντικά μετά την 8η Απριλίου. Από την άλλη μεριά, Έχουμε υποσχεθεί εμείς σε οικονομική βοήθεια ε, προς την Τουρκία. Ε, γνωρίζετε ότι υπάρχει η συμφωνία για το, ε, το 2016 και το 2007 να διατεθούν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που από την τουρκική πλευρά ε, ε, μας έχουν κατηγορήσει για καθυστέρηση διότι πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πώς θα δαπανηθούν οι πόροι αυτοί. Συνεργαζόμαστε κυρίως ε, με οργανισμούς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με το πρόγραμμα επισήτησης και την UNICEF. Ιδιαίτερα επικεντρωνόμαστε στην παροχή τροφίμων, την δημιουργία σχολείων, διότι ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι ε, ε, μέχρι 900.000 ε, παιδιά σχολικής ηλικίας βρίσκονται εκεί. Μία από τις συνέπειες της επίσκεψής μου ήταν ότι αποφασίσαμε να επενδύσουμε στην γλωσσική εκπαίδευση και των ενηλίκων, όχι μόνο των ε, παιδιών και νέων. Μέχρι και το 50% ε, κατά μερικού ε, των σύρων μεταναστών θέλουν να παραμείνουν στην περιοχή αυτή. Έτσι λοιπόν πέρα από την γλωσσική εκπαίδευση θα διαθέσουμε και πόρους ε, για ε, την ε, δημιουργία μικρών επιχειρήσεων και είμαστε διατεθειμένοι να διαθέσουμε πόρους για τις πόλεις και τα χωριά που έχουν υποστεί τις συνέπειες της μεταναστευτικής κρίσης και όπου έχει αυξηθεί δραματικά ο πληθυσμός λόγω της προσέλευσης μεταναστών. Υπάρχουν μέρη όπου έχει διπλασιαστεί ο πληθυσμός. Ε, είναι λοιπόν σημαντικό να προσέξουμε στα μέρη αυτά τις υποδομές. από τα 3 δισεκατομμύρια. Τα 2,2 προβλέπονται για προγράμματα και έργα συγκεκριμένα και από τα 2,27 δισεκατομμύρια μέχρι τώρα σχεδόν 700 εκατομμύρια ε, ε, έχουν αποτελέσει αντικείμενο συγκεκριμένων συμβάσεων και τα 180 εκατομμύρια έχουν ήδη διατεθεί. Έχουμε λοιπόν ε, εργαστεί πολύ καλά. Όσον αφορά την απελευθέρωση από τις θεωρήσεις, και εδώ στο Κοινοβούλιο και αλλού ε, έχουν συζητηθεί τα benchmarks, τα σημεία αναφοράς. εφαρμόζονται μέτρα στους διάφορους τομείς και το σημαντικότερο είναι η τροποποίηση της ε, νομοθεσίας ε, περί τρομοκρατίας ε, στην Τουρκία. Η Τουρκία μετά το πραξικόπημα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. υπάρχει πίεση χρόνου, αλλά τα σημεία σε αυτά, τα benchmarks, θα πρέπει να πληρούνται εντός λογικού ε, χρονικού διαστήματος, ώστε να μπορεί να υποβληθεί η θετική έκθεση. Και υπολογίζω αυτό να γίνει εντός του τελευταίου διμήνου του παρόντος έτους ώστε να μπορέσουμε και εμείς να δημοσιεύσουμε την ε, έκθεσή μας όπως έχουμε υποσχεθεί. Έχουμε λοιπόν αυτά τα 72 σημεία. στα οποία μένουμε. Από εκεί και πέρα όσον αφορά την ενέργεια, την οικονομία, έχουμε θετικές επαφές και συζητήσεις. Και όσον αφορά την Τελωνιακή Ένωση. Μέχρι τέλος της χρονιάς ε, θα έχει ολοκληρωθεί η εσωτερική αξιολόγηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη διαπραγματευτική εντολή. Γενικά λοιπόν ε, προοδεύουμε. Αλλά, όπως ήδη είπα, ε, το θέμα του κράτους δικαίου ανησυχεί όλους εμάς εδώ στο Κοινοβούλιο. Άλλωστε, σχετικά με τις ε, συλλήψεις που έχουν γίνει και δημοσιογράφων, ε, έχουν εκφραστεί ανησυχίες ε, από ευρωβουλευτές και εδώ και κατά την επίσκεψή μας στην Τουρκία. Προσωπικά βρίσκω θετικό ότι η Τουρκία δραστηριοποιείται περισσότερο τώρα στο θέμα της Συρίας. Αλλά τελικά και για την Συρία ισχύει αυτό που ισχύει για κάθε ένοπλη σύγκρουση, ότι θα επιδιώξουμε πολιτική λύση και όχι στρατιωτική. Είμαι πάντα αισιόδοξο Ε, είναι θετικό το θέμα της εκεχηρίας. Να προχωρήσω σύντομα ε, στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Ε, συνομιλήσαμε με την επικείμενη Εσθονική Προεδρία Ε, το 2017 ε, έχει προγραμματιστεί επί της αρχής ε, συνάντηση κορυφής για τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Και η Εστονία έχει προσφερθεί να οργανώσει τη διάσκεψη αυτή. Από ό,τι γνωρίζω μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Το αν δηλαδή αυτή η διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην Εστονία ή στις Βρυξέλλες. Δεν έχουμε αποφασίσει λοιπόν πού θα πραγματοποιηθεί. Έγινε ε, συζήτηση των Υπουργών Εξωτερικών στην Πρατισλάβα. Και εδώ υπόθηκε αυτό που πιστεύω και εγώ, ότι θα πρέπει να προσπαθούμε κάθε δύο χρόνια να έχουμε μια συνάντηση κορυφής, ε, αλλά να ε, αλλάξει η φύση των συναντήσεων αυτών, ε, να είναι συναντήσεις ε, για την εξέταση της κατάστασης, να γίνεται ένα stock-taking, διότι οι συναντήσεις κορυφής δημιουργούν προσδοκίες. Βλέπουμε τίτλους στις εφημερίδες, αλλά θέματα όπως η απελευθέρωση από τις βίζας ουσιαστικά έχουν αποφασιστεί. Τώρα βρισκόμαστε στην φάση της εφαρμογής. Θέλουμε λοιπόν ε, να έχουμε επίσημη συνεργασία. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα τέσσερα βασικά κεφάλαια στα, για τα οποία συμφωνήσαμε στη Ρήγα, δηλαδή κινητικότητα, ενίσχυση των θεσμών, καλή διακυβέρνηση, ε, Η κινητικότητα ε, έχει να κάνει και με τις επαφές μεταξύ ε, πολιτών, οικονομικές σχέσεις, διασυνδέσεις ανάμεσα στις χώρες της Ανατολικής Ιτωνίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν το καλοκαίρι, ε, συνάντηση των Υπουργών ε, Μεταφορών πραγματοποιήθηκε ε, μαζί με τους Υπουργού Μεταφορών των χωρών της Ανατολικής Γειτονίας και αποφασίστηκε η διεύρυνση του δικτύου του οδικού και του σιδηροδρομικού και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Τώρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και το ίδιο προβλέπεται σε άλλους τομείς με σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος Erasmus ε, ΣΥΝ, ώστε οι νέοι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να ε, έρχονται στην Ευρώπη και να σπουδάζουν. Στον τομέα των νέων ε, έχουμε και άλλα προγράμματα όπως είναι το Horizon 2020, Δημιουργική Ευρώπη, Κόσμε κλπ. Έτσι θέλουμε να ε, ε, έχουν οι χώρες αυτές πιο στενές σχέσεις με την Ευρώπη. Με μη δεσμευτικά νομοθετικά μέτρα να προωθήσουμε τη συνεργασία με την περιφέρεια αυτή και να φροντίσουμε έτσι να υπάρχει ε, σταθερότητα στην όλη περιφέρεια. Θα είμαι σύντομος όπως σας είπα. Όσον αφορά τον Νότο θα ήθελα να πω ότι σε σχέση με την Τινησία έχουμε αρκετά θετικές εξελίξεις. Ε, σε λίγες μέρες ε, θα ε, δημοσιεύσουμε την ανακοίνωση για την Τινησία. Σχεδόν διπλασιασμός του προϋπολογισμού προβλέπεται, 300, 300 εκατομμύρια προβλέπονται, όμως και η Τινησία θα πρέπει να συμβάλλει. Όπως και άλλοι, χαίρομαι και εγώ που η κυβερνητική κρίση της Άνοιξης κατέληξε θετικά με τη δημιουργία κυβέρνησης που είχε και την υποστήριξη της πλειοψηφίας στο Κοινοβούλιο. Και ελπίζουμε έτσι η χώρα να μπορεί να επικεντρωθεί περισσότερο στην πολιτική δουλειά. Στην Λιβύη δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά και εδώ βλέπω να υπάρχουν ε, τάσεις ε, προς σταθεροποίηση. Τον Οκτώβριο θα μεταβώ στην Αίγυπτο. όπου προχωρούμε αρκετά καλά στις διαπραγματεύσεις ε, για τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης με τη Ιορδανία και το Λίβανο. Ε, έχουμε ολοκληρώσει τις ε, εσωτερικές αξιολογήσεις ε, για τις συμφωνίες. Πρόκειται για δύο συμφωνίες οι οποίες θα συμβάλλουν σημαντικά στην βοήθεια προς τις χώρες αυτές για να αντιμετωπίσουν το μεταναστευτικό. Και τέλος, όσον αφορά την Παλαιστίνη, την χρήση των πόρων και τα διάφορα προγράμματα που παρακολουθούμε εκεί, όπως είναι τα, οι εγκαταστάσεις για αφαλάτωση στην ε, λωρίδα της Γάζας. Εάν δεν καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος μέχρι το 2020 να μην ε, υπάρχουν τέτοιες υποδομές και φανταστείτε τι σημαίνει αυτό για τη σταθερότητα και την ειρήνη στον τομέα. Ε, όσον αφορά τα, τις χώρες των ε, Δυτικών Βαλκανίων. Γενικά έχουμε θετικές εξελίξεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του, διάφορους ευρωβουλευτές ε, για τη δουλειά που έχουν κάνει σε διάφορες χώρες. Στην Αλβανία προβλέπεται δικαστική μεταρρύθμιση και θα είναι απαραίτητο να γίνει σωστή η εφαρμογή της μεταρρύθμισης αυτής. Ε, θέλουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε το μέσο της επιβράβευσης. Επίσης, ε, στην πρώην Ιουγκοσταβική Δημοκρατία της ε, Μακεδονίας Χωρίς πολύ θόρυβο, διαπιστώσαμε ότι τα πολιτικά κόμματα μπόρεσαν να συμφωνήσουν ε, πάνω σε ημερομηνία για τις εκλογές τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι πρέπει να εφαρμοστούν οι προτεραιότητες ε, στις μεταρρυθμίσεις. Ε, οι εκλογές δεν θα πρέπει να αποτελέσουν δικαιολογία, ούτε αποτελούν εκλογές στο τέλος της όλης συζήτησης. Ε, απαιτούνται ακόμα σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Όσον αφορά το κοσυφοπαίδιο, θα έχουμε τη δυνατότητα ε, να το συζητήσουμε αυτό. Ε, έχουν υπάρξει βήματα πρόοδου. Είναι όμως σημαντικό να έχουμε επανεκκίνηση του διαλόγου με την Σερβία. Μετά από διαπραγματεύσεις ε, μηνών. Ε, είναι θετικό σημάδι η ε, δημιουργία κυβέρνησης και η εκλογή Προέδρου. Σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε εκλογές στο Μαυροβούνιο. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και στη Βοσνία Ερσεγοβίνη έχουν υπάρξει βήματα προόδου, τα οποία θα πρέπει να αναγνωρίσουμε. και ελπίζω έτσι ε, να δοθεί η ορμή στην όλη διαδικασία. Επίσης, ε, χαίρομαι που ολοκλώθηκαν οι εκλογές ε, στην Κροατία. Το έθραυστο κλίμα στην περιφέρεια αυτή ελπίζουμε σιγά σιγά να μπορεί να, ε, να σταθεροποιηθεί. η συνάδελφος Πλέγκοβιτς θα με κοβήσει στις χώρες αυτές ε, και μέσα στις επόμενες εβδομάδες ε, θα δούμε ποιος ε, θα γίνει πρωθυπουργό. Όσον αφορά την διαδικασία των Δυτικών Βαλκανίων έχουμε καλή εξέλιξη, ωστόσο θα πρέπει να διασφαλίσουμε το αίσθημα οικειοποίησης στην περιφέρεια αυτή. για να διασφαλίσουμε την επιτυχία της διαδικασίας αυτές ε, στην ε, Λευκορωσία. Για την Λευκορωσία είχαμε μία πρώτη γνωμοδότηση πριν κάποιες εβδομάδες. Ε, υπάρχουν εδώ σημαντικά ελλείμματα όσον αφορά την δημοκρατία, αλλά χαιρόμαστε με κάθε εξέλιξη θετική που βλέπουμε. Μετά από 20 χρόνια είδαμε εκλογή δύο ανεξάρτητων ε, βουλευτών ε, στο Κοινοβούλιο. Στην ε, Γεωργία επίσης επικίνδυνε εκλογές. Και εδώ είναι σημαντικό να διατηρηθεί το ήρεμο κλίμα μέχρι το τέλος της διαδικασίας αυτής. Επίσης για την Αρμενία έχουμε κάποιες ανησυχίες, αλλά ελπίζουμε να, ε, έχουν, ε, να ε, συγκρατηθεί η κατάσταση εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Αλλά... Μια και θα χάσουμε έναν πολύτιμο αντιπρόεδρο που πρέπει να πάει σε μια άλλη συνεδρίαση με όλες τις διαδικασίες που πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα. Ας ξεκινήσω λοιπόν ε, πρόσφυγες. Αίγυπτος, Λιβύη. Πάνω από 100.000 λέει φτάσανε από τη Λιβύη στην Ιταλία. Θα πρέπει να υπάρχουν οι συνθήκες για να μην φτάνουμε αυτά τα άθλια φουσκωτά. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να συζητήσουμε τις αρχές της Λιβύης, της Αιγύπτου, γιατί μικρότερα λιμάνια της Δυτικής Αιγύπτου φαίνεται ότι χρησιμοποιούνται για να περάσουν. Αλλά ας ακούσουμε τον κύριο Πρέντα τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ευχαριστούμε που ήρθατε και μας ε, μιλήσατε με τέτοια πληρότητα και έχω κάποια παρατήρηση πολύ σύντομη. Όσον αφορά την Τουρκία, όλοι έχουμε καταδικάσει το πραξικόπημα. Αυτά που συμβαίνουν μετά το πραξικόπημα είναι πάρα πολύ ενσχυτικά ακριβώ σε σχέση με αυτά που είχαμε συζητήσει και πριν το πραξικόπημα, δηλαδή για τον ορισμό τη τρομοκρατία. Γιατί η μεγάλη εμπλοκή που έχει επελθεί όσον αφορά το θέμα τη απελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίων είναι ο ορισμό τη άγκυρα για την τρομοκρατία και ακριβώς μετά το πραξικόπημα ορίζει ως τρομοκράτες τους εχθρούς του Ερντογάν. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα και θεωρώ ότι η κρίση είναι πάρα πολύ σοβαρή, αφορά τον πολιτικό μας διάλογο και θα πρέπει αυτό να αναγνωριστεί. Γιατί ταυτόχρονα λέει ο Ερντογάν ότι αν δεν απελευθερώσετε τις ε, βίζες τότε θα μπλοκάρουμε τη συμφωνία για τους ε, μετανάστες. Άρα γι' αυτό σας λέω ότι εδώ πέρα έχουμε μεγάλη κρίση όσον αφορά τον ε, πολιτικό διάλογο σχεδόν η μισή ήταν την αντιπολίτευση για την ηλεκτροκρασία ε, αλλά οι περισσότεροι τελικά που ε, ε, εξελέγησαν νομίζω ότι μιλάγαμε τα τελευταία χρόνια για πλουραλισμό με, με ένα με μονοκομματισμό ταυτόχρονα τώρα κάτι άλλο μια που ο πρόεδρος της υπερδινιστερίας είπε ότι θέλει να προσχωρήσει στην Ρωσία επί τη βάση του δημοψηφίσματος που έγινε πριν από 10 χρόνια. Άρα προσοχή σε αυτή τη νέα κρίση. Ευχαριστώ να μας πείτε και δύο λόγια για την Βοσνία και για το σχετικό δημοψήφισμα. Ευχαριστώ για την κατανοησή σα, Πρόεδρε. Πρόεδρος. Εκτός μικροφώνου. Κυρία Πύρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, νομίζω είναι πάρα πολύ αξιόλογο το ότι εσεί και η Φεδερικά Μογγερίνη πήγατε στην Άγγελ την περασμένη ε, εβδομάδα και συνεχίστηκε ε, ο πολιτικό διάλογο υψηλού επίπεδου. Είναι κάτι το οποίο χρειαζόταν πάρα πολύ. Γιατί βέβαια δεν συμφωνούμε πάντοτε σε όλα. Και με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι αύριο στην Ολομέλεια θα υπάρξει εντελή συζήτηση. Κάτι άλλο για την Τουρκία. Πέστε μας Δύο λόγια όσον αφορά ε, τις ε, βίζες θα ε, δημοσιοποιήσει μια έκθεση η Ευρωπαϊκή Τροπή. Έχει υπάρξει κάποια συγκεκριμένη συμφωνία στον πρώτο ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης σε σχέση με την υποστήριξη, σε σχέση με την εποπτεία και παρακολούθηση. Τότε που πήγατε είδατε ότι είχαμε 40.000 δάσκαλους και διδάσκοντες που με τον ισχυρισμό για την κατηγορία ε, συνελήφθησαν ότι είχαν σχέση με το ΠΚΚ και χθε είχαμε 28 δημάρχους επίσης οι οποίοι συνελήφθησαν. Βλέπουμε ότι η κατάσταση της ανάγκης τώρα χρησιμοποιείται και έναντι άλλων και όχι μόνο έναντι των προεξομεδιών. Για πετε μας, πώς βλέπετε αυτές τις εξελίξεις. Τώρα, τελευταία ερώτηση όσον αφορά τη Συμφωνία Ένωσης και Τουρκίας. Μία από τις δικές μας υποσχέσεις ως Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από το άνοιγμα των κεφαλαίων, πέρα από τις χρηματοδοτήσεις, ήταν ότι θα υπάρξει μεγάλη έκταση σε επανεγκατάσταση και μετεγκατάσταση των ε, Σύρων. Και οι 28 ε, μετέφεραν χίλιους από την Τουρκία ή στην Ευρώπη. Πρόκειται να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση τις αμέσως επόμενες ημέρες. <laughs> You might guess. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για την εισήγησή σας. Ήθελα να σας πω κάτι για την πλατφόρμα της ε, γειτνίασης προς Ανατολάς. Είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, έχει μετασχηματίσει πολλές χώρες και έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Πόσο βαθιές μεταρρυθμίσεις έγιναν, αλλά και ακόμα βέβαια θα πρέπει να γίνουν, να έχουμε καλύτερη ποιότητα σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις και τελικά να μπορέσουμε να αποκομίσουμε τα αποτελέσματα τα οποία προσδοκούμε. Όμως κάποιες χώρες βρίσκονται ακόμα σε μια ενδιάμεση κατάσταση πρέπει να επιδείξουν ε, υπομονή αλλά τι θα γίνει με τις χώρες οι οποίες δεν μπαίνουν στην πλατφόρμα της ε, εταιρική σχέσης προς Ανατολάς. Ας πούμε έχουμε τον Κάφκαζο. Ε, Ανατολική Ευρώπη γίνανε κάποιες εκλογές και ο στην εκθεσή του λέει ότι τα πρότυπα του ΩΣΑ δεν πληρούν το είδαμε τις ε, κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας αλλά δεν βλέπουν να υπάρχει καμία αντίδραση. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα περιμέναμε. Άρα τι λέτε για αυτές τις χώρες, εκείνες ε, οι οποίες ε, δεν είναι σε τέτοιο επίπεδο ούτω ώστε να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της γητρικής σχέσης προς Ανατολάς ούτω ώστε να μπορέσουν να αποκομίσουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, εμείς θα πρέπει να είμαστε σκληροί. Θα πρέπει να τηρήσουμε τις προποθέσει που έχουμε τάξει. Να τηρούνται τα συμπεφωνημένα. Για το καλό των χωρών αυτών. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτούς τους κακούς μαθητές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε και εγώ έχω κάποιες ερωτησούλες όσον αφορά την ε, σχέση εταιρικής σχέσης προς Ανατολάς, την πλατφόρμα μάλλον εταιρικής σχέσης και πιστεύω ότι το πιο οξύ πρόβλημα τώρα είναι το εξή. Τι γίνεται με Γεωργία και Ουκρανία όσον αφορά την κατάργηση της βίζα των διαβατήριων. Φυσικά και θα γνωρίζετε ότι πήγε καλά η διαδικασία η κοινοβουλευτική και οι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ κάνανε ό,τι έπρεπε και πάει το θέμα για ολομέλεια. Όμω, τι γίνεται στο Συμβούλιο, τι γίνεται με τι ε, επιφυλάξει. Βασίζονται σε κάποια γερά επιχειρήματα ή απλώ είναι δισταγμό και φόβο για το πολιτικό κλίμα, για τη στάση τη Γερμανία κλπ. Τι γίνεται με αυτέ τι ρήτρε διαφύλαξη που τώρα συζητούνται, πώ το βλέπετε εσεί, τι προτείνετε, τι νομίζετε ότι θα συμβεί. Επίσης, κατά δεύτερο λόγο ή για τη Λευκορωσία. Ίσως είναι πρόημο να πούμε ότι έχει λιώσει ο πάγος, αλλά έχουμε την εκλογή κάποιων μέλων της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι ένα βηματάκι. Καλό. Άρα θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση με τα θα γίνουν, αλλά βέβαια και θα πρέπει οι εκλογές να ζηγιστούν επί τη βάση των συστάσεων του ΟΣΑ, όπως είχαν διατυπωθεί αυτέ μετά τι ε, προεδρικές εκλογέ, κατά τρίτο λόγο, το Αζερβαϊτζάν. Είπατε ότι είχαμε κάποια αντιπροσωπεία που μετά από, μεγάλη, μετά από πολύ και μετά μεγάλη διακοπή των επισκέψεων εκεί θα ταξιδέψει την επόμενη εβδομάδα εκεί και πρόκειται επομένω για ένα δημοψήφισμα που θα γίνει 25 ή 26 του τρέχοντος μηνός. Τι λέει η Επιτροπή για αυτό το δημοψήφισμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ και εσά που είχατε την καλοσύνη να έρθετε σήμερα εδώ και να μα ενημερώσετε για όλα αυτά τα θέματα που έχουν σχέση με τι χώρε τη περιφέρεια. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στην Τουρκία. Αν ε, κάποιο είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί τι εδώ συναντήσει, ε, θα έβλεπε ότι αναμασούμε τα ίδια πράγματα. Η Τουρκία ουδέποτε στην πραγματικότητα ήταν μια δημοκρατική χώρα. Τώρα, μετά την ε, διενέργεια του πραξικοπήματος, ο Ερντογάν βρήκε ευκαιρία να καταλύσει όποια προσχήματα τηρούσε δημοκρατικά για να μπορέσει να κυνηγήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Από την άλλη πλευρά, εμείς βλέπουμε πρόοδο. Και ενώ έχουμε την μεγάλη ευκαιρία να πιέσουμε την Τουρκία, επιτέλους να φανεί συνεπίση στις υποχρεώσει που έχει απέναντι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κάνουμε, βλέπουμε ότι και πιστεύουμε ότι η Τουρκία θα τηρήσει τι υψηλέ ε, προδιαγραφέ και τα πρότυπα στα οποία αναφερθήκατε, ότι θα υπάρξει διαφάνεια, θα σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλα αυτά τα ωραία. Μεγάλε προσδοκίε, όπω έλεγε και ο Κάρλο Δίκεν. Αυτό όμω μπορούσε να το πει. Εμεί δεν μπορούμε να το πούμε. Γιατί ζούμε την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα μα δίνει να αντιληφθούμε ότι εάν συνεχίσουμε με αυτή την πολιτική δεν πρόκειται ποτέ να βρούμε άκρη με την Τουρκία. Ήδη έχει αρχίσει και αυξάνει τις ροές των παρανόμων μεταναστών προς τα ελληνικά νησιά. Και επειδή δεν θέλω να μακρηγορήσω, τελειώνω λέγοντας το εξής. Είπατε, είπατε ότι βλέπετε πρόοδο και είναι θετικό το γεγονός ότι η Τουρκία εισέβαλε στη Συρία. Έκανε δηλαδή αυτό που έκανε πριν 40 χρόνια και στην Κύπρο. Και αυτό για εσά είναι θετικό. Επειδή λοιπόν ξεφεύγει από τη δική μου λογική, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μου το αναλύσετε αυτό το πράγμα. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε εισβολή στρατιωτική σε μια γειτονική χώρα και αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Και, και, και τέλος, πώς είναι δυνατόν να περιμένουμε πολιτική λύση όταν έχουμε στρατιωτική εισβολή. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα πρώτα θα ήθελα να σας πω για τα αποτελέσματα των εκλογών στην Λευκορωσία. Γνωρίζω τη χώρα και έχω ταξιδέψει τέσσερις φορές για να επισκεφθώ τη χώρα. Και έχω συνεχή επαφή με τους δημοκρατικούς φορείς. Πιστεύω ότι έχουμε δύο μέλη της που εξελέγησαν ότι είναι ένα πάρα πολύ μικρό βήμα πρόοδου. Έκανε πάρα πολλά Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρα πολλά μηνύματα έχουμε στείλει στη χώρα. Δεν αρκεί αυτό το οποίο έγινε. Άρα θα πρέπει να ε, το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Πώς θα προχωρήσουμε όσον αφορά τον διάλογο. Και το διάλογος είναι μεγάλη υπόθεση που το λέμε αυτό. Γιατί μιλάμε για μετασχηματισμό προς μια δημοκρατική κοινωνία στη χώρα. Ε, επίσης θα συμφωνήσω αυτήν την συνάντηση κορυφής της εταιρική σχέσης προς Ανατολάς. Stock taking όπως και το είπατε γιατί έχουμε. Τα γεγονότα στην Ανατολική Ευρώπη, έχουμε το μεταναστευτικό. Όλα αυτά έχουν ε, σκιάσει αυτήν την υπόθεση, έχουν κάνει τη φλόγα της να τρεμοσβήνει. Αλλά πρέπει, πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση ψηλού επίπεδου. Ο επόμενος. Κύριε Κύριε Επίτροπε, καλύπτεται ένα χώρο που είναι μεγαλύτερος και από την ίδια την Ευρώπη. Όμως υπάρχει έλλειμμα αναλύσεως στο τι συμβαίνει, τι εξελίσσεται σε αυτόν τον χώρο, σε αυτήν την περιοχή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και Ευρώπης. Εμείς στο γόνατο νομίζω λαμβάνουμε τις πολιτικές ε, αποφάσεις για διάφορες ε, χώρες, περιπτωσιολογικά. Και η προσέγγιση στις χώρες της εταιρικής σχέσης προς Ανατολάς νομίζω ότι έχει θαμπόσει. Άρα ας εστιάσουμε την προσοχή μας σε κάποια στοιχειώδη βασικά σημεία. Ας πούμε την ανάπτυξη δημοκρατικών θεσμών. Επίσης, άλλο έλλειμμα στο επίπεδο της ανάλυσης υπάρχει το οποίο διαπιστώνω. Οπότε, αν θέλουμε να διαμετρήσουμε κάποιον ρόλο σε όλη αυτή την περιοχή, θα πρέπει να κάνουμε μια αξιόπιστη ανάλυση για το τι πρόκειται να γίνει την επαύριο στις χώρες αυτές που μας απασχολούν. Επίσης, έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Είστε από τους λίγους πολιτικούς, αλλά και ο πρόεδρος μας, πήγε, που πήγατε στην ε, Τουρκία, αλλά δεν έγιναν αρκετές επαφές μετά από το γεγονότα του προεξκοπήματος. Ακόμη δεν έχουμε κατανοήσει το τι έγινε εκεί. Τι είναι το φαινόμενο Γκιουλέν, ποια είναι η σημασία του, ποια είναι η σημασία του για μας σήμερα. Επίσης, ο Ερντογάν διώγει τους Γιουλενιστές παντού. Και υπάρχουν πράκτορες του Ερντογάν και στις δικές μας χώρες που αναζητούν τους Γιουλενιστές, Ασκούν πίεση στις κυβερνήσεις των χωρών μας. Άρα, θα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο για να καταλάβουμε τι γίνεται στην Τουρκία και να καταλάβουμε τι προσδοκά από την Ευρωπαϊκή Ένωση η χώρα αυτή. Και σας ευχαριστώ. Ήσασταν πολύ γενναιόδος πρόεδρε αυτή τη φορά. Ευχαριστώ. I don't hear what you say, Δεν άκουσα τι είπατε πρόεδρε κ. Μπουτικόφερ γιατί μίλησε εκτός μικροφώνου ο πρόεδρος. Θα ήθελα ξεκινώντας να κάνω μια εισαγωγική παρατήρηση στον Επίτροπο για την Τουρκία. Είπατε ότι όλοι κατεδίκασαν αμέσω την απόπειρα του πραξικόπηματος. Ωστόσο πρέπει να ομολογήσουμε ότι η αλληλεγγύη, ο βαθμός αλληλεγγύη που εκδηλώθηκε έναντι της ε, Τουρκίας την ώρα που εκδηλώθηκε το πραξικόπημα ήταν ελλειπή. ένα μόνο Ε, πολιτικός από την Ευρώπη ε, πήγε γρήγορα στην ε, Τουρκία για να εκδηλώσει υποστήριξη και αυτή είναι η Βρετανή Πρωθυπουργό. Ήταν κακό δείγμα πολιτικής από πλευρά της Ευρώπης και νομίζω ότι αυτή την αμέλεια να μην την αγνοήσουμε, δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε ελαφρότητα. Επίσης θα ήθελα ιδιαίτερα να σημειώσω και να ρωτήσω πώς ε, κρίνετε εσείς την αντιμετώπιση του HTP, του κόμματος της αντιπολίτευσης, που δεν εκλήθη να συμμετάσχει σε κοινέ ε, ε, δράσεις. Ερωτώ λοιπόν πώς κρίνεται αυτή την τελευταία κλιμάκωση. Και επίσης η επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων στους προσαρατολάς Πώς θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει, δηλαδή το κεκτημένο των ε, διαδικασιών και κανόνων για τους διαγωνισμούς θα, θα επεκταθεί και σε αυτές τις χώρες. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, ήσασταν στη Σερβία την προηγούμενη εβδομάδα. Διάβασα και σε ένα ανακοινωθέν τύπο ότι παρακολουθήσατε και συνεδρίαση κυβερνητικού συμβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν ε, να διατυπώσω τις εξής ερωτήσεις. Ο Πρωθυπουργό σας εξέθεσε ή αναφέρθηκε στο πρόγραμμα το κυβερνητικό για τα επόμενα χρόνια εν ώψη των ε, μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για, τα, για την προσαρμογή στα κεφάλαια 23 και 25 και επίσης μετά τις εκλογές 11 Σεπτεμβρίου. Πώς νομίζετε ότι θα συνεχιστεί η κατάσταση στη Σερβία. Ήτανε δυσμενής πιστεύω η κατάσταση τους τελευταίους μήνες. Ήταν πολύ αρνητική η ρητορική της κλιμάκωσης. Νομίζετε ότι θα έρθει η ώρα σύντομα να γίνονται ε, προεκλογικές εκστρατείες χωρίς εθνικισμούς και κλιμάκωση. Κυρία Λούνατσεκ, πρόεδρε, ερώτηση για Τουρκία καταρχάς και για τα Βαλκανικά μετά, τα Βαλκανικά κράτη. Πώς θα αντιμετωπίσει το Συμβούλιο περαιτέρω την ε, Τουρκία. Ξέρετε ότι έχουμε μεγάλη σύντηση και στην Αυστρία. Η κυβέρνηση της Αυστρίας είπε ότι θέλει να, διακόψει τις, να διακοπούν οι διαπραγματεύσεις. έχετε θέματα της διεύρυνσης βεβαίως της αρμοδιότητές σας. Πώς βλέπει τα πράγματα η Επιτροπή και πώς ε, σκοπεύει να τοποθετηθεί στην επερχόμενη σύνοδο. Νομίζω ότι δεν είναι εύστοχη η διακοπή των συνομιλιών. Αν και βεβαίω θα πρέπει να προσαρμοστεί ή θα πρέπει να περάσει πολλή χρόνο και να προσαρμοστεί η κατάσταση στα νέα δεδομένα για να ξαναρχίσουν οι συνομιλίε. Ε, με το HTTP, με εκείνου ε, από τα μέσα μαζική ενημέρωση που μπορεί να μην έχουν ε, χάσει τη δουλειά του ή να μην βρίσκονται στη φυλακή. Έχετε επικοινωνία χωρίς να ανήκουν βέβαια στην κυβέρνηση αυτή, και για τα Βαλκάνια. Και δεν θα είναι το κοσμοπέδιο το θέμα μου σήμερα, αλλά ε, η Αλβανία, σχετικό, ενεργειακά σχέδια, ανέγερση ενεργειακών σταθμ, σταθμών παραγωγής ενέργειας, ιόκα, πώς μπορεί η Επιτροπή να παρακολουθήσει έργα τα οποία δεν αναπτύσσονται με βάση τα ευρωπαϊκά κριτήρια ή πώς μπορεί η Επιτροπή, πώς μπορείτε εσείς να εξασφαλίσετε την τήρηση των ευρωπαϊκών κριτηρίων. Τελευταία, η Βοσνία. Η Ρεπούμπλικα Σέρψκα έχει προβλέψει, έχει προσδιορίσει για την 20η Σεπτεμβρίου ένα δημοψήφισμα με επέτειο της διακηρύξεως του Κάρασιτς ε, του 1992. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Ρωτώ λοιπόν τι νομίζετε ότι μπορούμε να κάνουμε, τι σκοπεύετε να κάνετε εσείς, ε, βέβαια πάντα με την ελπίδα ότι δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά αυτή η εκδήλωση και δεν θα ενισχυθούν οι εθνικιστικές ε, και ακραίε δυνάμεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συνεχίσω λίγο στα όσα είπε ο αξιότιμο εδώ γείτονο μα του στον Μακαλιστεριά, γιατί μα προβληματιζόμαστε πάρα πολύ όσον αφορά τι πολιτικέ διμερεί σχέσει μεταξύ Κροατία και Σερβία. Γιατί τα πράγματα δεν είναι και τόσο τέλεια, τόσο ειρηνικά, τόσο θετικά, τόσο επικοδομητικά, για να το πω έτσι διπλωματικά. Και ε, ξέρετε ε, τι θέση υιοθέτησε η Σερβία και νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση είναι το να μην υπάρξει απάντηση. Και τώρα υπάρχουν ε, κάποιες φήμες ότι η καινούργια κυβέρνηση, η πιο θετική θέση, εγώ θα ήμουν τόσο αισιόδοξο. Μπορείτε να μου πείτε δύο λέξεις πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια σύντομη ερώτηση. Η κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο μέχρι τώρα ήταν καταστροφική. Ένα-δύο παραδείγματα. Έξι εκτελέσεις για αδικήματα που δεν θα μπορούσαν καν να έχουν διαπράξει οι κατηγορούμενοι γιατί ήταν στη φυλακή την εποχή που διαπράγησαν. Και παρόλα αυτά ε, εκτελέστηκαν. Επίσης η κατάσταση παραμένει ε, όπως είχε γιατί οι τελευταίες συντήσεις δεν έχουμε λάβει. Και Δεύτερη ερώτηση, σε τέτοιες περιπτώσεις πώς δράει η Επιτροπή. Σας ευχαριστώ για την Τουρκία και πάλι. Αυτά τα οποία δεν είδαμε στη συνολική εικόνα και που είδα στις συνομιλίες με Τούρκους ήταν το πόσο πόσο είχε διεισδύσει στο κράτος το κίνημα Γκιουλέν στη δικαιοσύνη, στην αστυνομία, στις αρχές της, ε, της τάξης, στην εκπαίδευση. και παρατρίχα γλιτώσαμε το πραξικόπημα. Σε πολλές συνομιλίες που είχα εκεί διαπίστωσα πολύ έντονη συγκινησιακή φόρτιση. Κάποιοι μάλιστα είχαν ε, για ελάχιστο γλιτώσει από κίνδυνο ζωής από αυτό το πραξικόπημα. Και αυτό επηρεάζει ακόμη τις αντιδράσεις τους, τον τρόπο με τον οποίο μιλάνε. Νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουμε, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αξιολογήσει κανείς ποια θα έπρεπε να είναι η κατάλληλη και απαραίτητη αντίδραση για το πραξικόπημα. και πώς μπορεί ενδεχομένως να έχει γίνει υπέρβαση των συνθήκων μιας κατάστασης ανάγκης προκειμένου να εκμεταλλευτεί κανείς την κατάσταση και να επιτύχει άλλους στόχους. Είναι και αυτό κάτι πρέπει να αξιολογήσουμε σύντο χρόνο. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη. για την έκθεση σχετική με την απελευθέρωση από την υποχρέωση θεώρηση των διαβατηρίων. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη η ημερομηνία, δεν υπάρχει προθεσμία, διότι αυτό θα εξαρτηθεί από την τήρηση των προποθέσεων από πλευρά τη Τουρκία. Και σε αυτό δεν μπορώ να δώσω πιο συγκεκριμένη απάντηση. Ο Ιούνκερ, ο Τούσκ, στο πλαίσιο τη Συνόδου Κορυφή G20, το επιβεβαίωσαν, έχει επιβεβαιωθεί επανειλημμένο εξάλλου και πρέπει να ε, βρεθεί μια λύση, το δέχεται και η Τουρκία αυτό. Και εν προκειμένου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης μπορεί να βοηθήσει ώστε να απαλληφθούν κάποιες παρεξηγήσεις. Εμείς ως Επιτροπή δεν παραπέμψαμε το θέμα στο Ευρω... Συμβούλιο της Ευρώπης. Απλώς αξιοποιούμε την ε, τεχνογνωσία του, τις ειδικέ του γνώσεις και την πολιτική αξιολόγηση της κατάστασης από πλευρά του Συμβουλίου της Ευρώπης. για την κυρία Λούνατσεκ, τον κύριο Μπιουτικόφερ και άλλους ε, που έθεσαν το σχετικό ερώτημα. Εγώ στις, σε επισκέψεις μου συναντώ και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Ήμασταν μόνο για κάτι λιγότερο από μια μέρα εκεί, επομένως ε, δεν είχαμε τόσο χρόνο, αλλά συναντηθήκαμε και η κυρία Μογκερίνη και εγώ με τέσσερα πολιτικά κόμματα. Το συντηρητικό εθνικιστικό κόμμα ε, MHP, το CHP, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και το HTP. Και βεβαίως ε, ήμασταν και στο, στην έδρα του AKP. Με μεγάλη προσοχή να μην παρεξηγηθεί καμιά κίνηση βέβαια. Ε, εγώ είχα ανέκαθεν την γνώμη και έχω επισημάνει στους Τουρκούς συνομιλητές ότι θα ήταν ε, καλό το HTP ως πολιτικό σκέλος του κουρδικού κινήματος να ενισχυθεί. Αλλά βέβαια αυτό απαιτεί ταυτόχρονα και το HTP να ε, κρατήσει σαφείς αποστάσεις από το PKK, από το PKK και να καταδικάσει η αδίποτε μορφή βίας. Ε, και για να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν βλέπουμε τέτοιες σαφείς αποστάσεις και καταδίκη. Το HDP μπορεί να καταδικάσει ενδεχομένως ή να απορρίψει τη βία κατά πολιτών μόνο, αλλά σε αυτό δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε μαζί τους γιατί η βία είναι βία και είναι πάντοτε καταδικαστέα. Εδώ λοιπόν χρειαζόμαστε πιο σαφείς τοποθετήσεις από πλευράς του HDP. Αλλά όπως είπα και πριν, το HTTP είναι για μένα η πρώτη πρόσφορη βάση για μια πολιτική λύση. Αλλά όπως είπα, πρέπει να δούμε σαφείς τοποθετήσεις για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και παρερμηνίες Για το όλο ζήτημα της ε, απαλλαγής από την υποχρέωση των ε, διαβατηρίων εδώ Εκκρεμούν τα ζητήματα της Ουκρανίας, της Γεωργίας, στη συνέχεια βέβαια του και της Τουρκίας σε σχέση με τα προβλήματα λοιπόν αυτά, με τα ζητήματα αυτά και εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήθελα να σα επισημάνω πω ακολουθούμε μια ω ε, το δυνατόν πιο αντικειμενικά οργανωμένη μεθοδολογία με συγκεκριμένα ορόσημα, benchmarks, σε συνεργασία με τους εταίρους, σε ε, συνομιλίε διαρκή και με το Συμβούλιο και όταν τηρούνται αυτά τα ορόσημα θα ήταν ζήτημα αμφισβήτησης της μα μας αξιοπιστίας. των μην εγγυηθούμε την ε, απελευθέρωση αυτή από την υποχρέωση θεώρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ήπια δύναμη. Και ως εκ τούτου, αφού δεν θα μπορούσαμε να ασκήσουμε βία ή με δύο τρόπο να επιβάλλουμε την ισχύ μας, η ισχύ μας είναι η αξιοπιστία μας η τήρηση των κανόνων και πάνω απ' όλα τήρηση των δικών μας κανόνων, αυτών που εμείς έχουμε ορίσει. Γι' αυτό και ιδιαίτερο θέλω να τονίσω που σε σχέση με τους εταίρους πρέπει να είναι ε, σίγουροι ότι όταν τηρούνται οι κανόνες, ε, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο πάντα. Αλλά βεβαίως υπάρχουν άλλα ζητήματα πολιτικής επιλογής, η επέκταση της λεγόμενης ρήτρα ασφαλείας, διασφαλιστικής δικλίδας, Πρόκειται για ένα ζήτημα θεσμικό που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και αφορά την επιλογή της ε, κατεξουσιοδότησης της εφαρμοστικής πράξης. Ε, εγώ θα ήθελα να απευθύνω έκκληση να επιληθεί το ταχύτερο δυνατό το πρόβλημα αυτό, γιατί ε, με όλη την σημασία του βεβαίως, από αυτό το θέμα εξαρτάται η πρόοδος της υπόθεσης της απελευθέρωσης από την υποχρέωση των διαβατηρίων για τα κράτη αυτά. Εκ μέρους μου λοιπόν δεν βλέπω επί της ουσίας προβλήματα, αλλά βλέπω να σταματάει η συζήτηση σε ένα θεσμικό πρόβλημα. εδώ, ιδιαίτερα για την Ουκρανία και την Γεωργία, νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να αποστολούν τα κατάλληλα πολιτικά μηνύματα πάνω απ' όλα ότι τηρούμε τους κανόνες που έχουμε εμείς οι ίδιοι ορίσει. Για τη Ρωσία δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένο από τη ε, βαθμό των εξελίξεων που εμείς τουλάχιστον επιδιώκαμε. Από πλευράς ε, διορθώνω. Ε, θα πρέπει πιστεύω να δούμε, να περιμένουμε να δούμε βήματα από πλευράς Λευκορωσίας που θα ε, αποτελούν αντανάκλαση της καλής βούλησης που δείξαμε εμείς από πλευράς μας. Και έτσι θα μπορούσαμε και από ευρωπαϊκής πλευράς να λάβουμε τις ε, κατάλληλες αποφάσεις. για, την, ε, για τις τελευταίες ερωτήσεις, για το αν θα πρέπει να αυτοσχεδιάζουμε και ποτέ ποτέ. Βεβαίως αναγκαζόμαστε να αυτοσχεδιάζουμε όταν ε, βλέπουμε εξελίξεις τις οποίες δεν είχαμε μπορέσει να προβλέψουμε πριν. Ε, πάντως από πλευρά μου, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πως υπάρχει μια σταθερή γραμμή, μια γενική γραμμή. Η γενική αυτή γραμμή είναι σταθεροποίηση στην γειτονία μας. Βεβαίως αυτό θα πρέπει να το χειριστούμε με μια ευελιξία, πράγμα το οποίο σημαίνει ποτέ ποτέ και αυτοσχεδιασμό, αλλά ο στόχος, η γενική γραμμή είναι σταθεροποίηση. Σταθεροποίηση μπορούμε με τα δικά μας μέσα και τις δυνατότητές μας να εξασφαλίσουμε μόνο εφόσον υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, εφόσον μπορούμε να βοηθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη να προχωρήσει μαζί με το κράτος δικαίου. Σε ορισμένα από αυτά κράτη δεν έχουμε τόση μεγάλη ευχαίρεια να υποστηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών, διότι υπάρχουν τάσεις ε, την οικονομική υποστήριξη να μην επιτρέπουν να την διαχειρίζονται ξένες οργανώσεις ή να μην τίνουν να επιτρέπουν να τη διαχειρίζονται ξένες οργανώσεις. Αυτό είναι κάτι πρέπει να συζητούμε πάντα με τους εταίρους. Αυτό είναι ένα ζήτημα, παραδείγματι, με την Αίγυπτο. Δεν μπορώ να σας πω ποιες είναι οι πιο πρόσφατες εξελίξεις σχέση με το ερώτημά σας, αλλά μπορώ να σας πω πως στις συνομιλίες μας με τον Τούρκο λέει ο μιλητής τώρα συνομιλητή μα. τα ζητήματα του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σημαντικό κομμάτι της συζήτησης για την ανάπτυξη των προτεραιοτήτων για την εταιρική σχέση που θέλουμε βέβαια να περιλάβουμε. Δυτικά Βαλκάνια. δυστυχώς σε σχέση με την ε, ειρήνευση βλέπουμε ότι οι επερχόμενες προεδρικές εκλογές στη Σερβία έχουν οδηγήσει σε μια όξυνση της ε, ρητορική που μετέρχονται οι διάφοροι υποψήφοι. Μάλλον ε, το αντίθετο από συμφιλιωτικές τάσεις βλέπουμε και μας ανησυχεί βεβαίως αυτό. Ε, έχουμε μπορέσει κάποιοι από εμά να κρατήσουμε στο δυνατόν χαμηλούς τους τόνους σε σχέση με ε, προκλήσεις στην Κροατία, κινήματα εκλογικά, να μην ε, οδηγήσουν δηλαδή σε ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση στη Σερβία. Αλλά θα χρειαστεί αυτοσυγκράτηση από κάθε πλευρά. Και θα πρέπει να υπάρξουν και από την άλλη πλευρά αντιδράσεις και προκλήσεις. Πάντα είμαι αισιόδοξο, αλλά αυτή τη φορά είναι περιορισμένη σε κάποιο βαθμό η αισιοδοξία μου. Πάντως νομίζω ότι μπορούμε να δράσουμε με ευφύ τρόπο και να κοιτάξουμε στο πρώτο τρίμηνο που έχουμε μια συνάντηση των αρχικών ε, κρατών και κυβερνήσεων των Δυτικών Βαλκανίων και όπου θα ήθελα να είμαι σε θέση να προσκαλέσω τον νέο Πρωθυπουργό της Σερβίας, ε, θα έθετα, εφόσον έχω αυτή τη δυνατότητα, το ζήτημα του εθνικισμού, των λαϊκισμών, στην περιοχή αυτή που πρέπει κατά προτεραιότητα ε, να συζητηθούν. Και πρέπει νομίζω να συζητήσουμε εν όλο το ζήτημα του τι μπορούμε εμείς να κάνουμε, τι μπορούμε να προσφέρουμε. Για τη Βοσνία. Σύντομα. Γιατί έχω συνομιλήσει πολύ και με τον Βούτσιτς, και έχει επηρεάσει και το Τούντικ. Αν δείτε τις τελευταίες του δηλώσεις αυτό το Σαββατοκύριακο. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και με τάση συμφιλιωτική μια δήλωση του ε, ακυρωτικού δικαστηρίου της Βοσνίας Ερζεγοβίνης που δεν, ακυρ, δεν ανακαλεί, δεν ακυρώνει την απόφαση του δικαστηρίου αλλά τουλάχιστον ε, καλεί την ε, Ρεπούμπλικα Σέρψκα να μην πραγματοποιήσει το δημοψήφισμα. ελπίζω ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει μια θετική εξέλιξη για την κυρία Λούνασεκ και την Αλβανία. Δεν έχω συγκεκριμένη απάντηση να σας δώσω αυτή τη στιγμή, μόνο καταρχήν θέλω να σημειώσω πως ε, με δική μου πρωτοβουλία έχουμε αναπτύξει ένα master plan για τα Βαλκάνια και την ενέργεια, ιδιαίτερα τα ύδατα και βλέπουμε ότι δεν αξιοποιούνται επαρκώς ως ενεργειακή πηγή τα ύδατα στα Βαλκάνια αλλά και ιδιαίτερα την Αλβανία. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι και για λόγους περιβαλλοντικούς πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη ενεργέτερο ιδιαίτερο βάρο σε αυτή την πτυχή. Ο κύριο Πίβαλξ, ο αρμόδιο επίτροπο, μου είχε πει ότι η Δυτική η Βαλκανική θα μπορούσε να είναι ανεξάρτητη, αυτόνομη ενεργειακά, αν αξιοποιούσε επαρκώ όλου τους ενεργειακού πόρους που διαθέτει. Αυτό έχει τεράστια πολιτική διάσταση και από αυτή τη ενία είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αμελήσουμε, να παραμελήσουμε. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συζητήσουμε όλα τα θέματα και τώρα, εάν ε, νομίζετε και ότι έχω καλύψει όλα τα ζητήματα, να μην μείνω εγώ το τελευταίο εμπόδιο στο δείπνο σας. Α, τη δική μου την, απα... την ερώτηση δεν την απαντήσατε. Τι Λιβύη, πρόεδρε, πώς το ξέχασα. Εν όλων, λοιπόν, μπορούμε να διαπιστώσουμε. Αυτό, ξέρετε, με το μισογεμάτο και μισοάδιο ποτήρι, ότι οι πρόσφυγες ε, από τη Δυτική Μεσόγειο μπορεί να μην μειώθηκαν, αλλά πάντως δεν αυξήθηκαν το τελευταίο έτος. Είναι κατά το ίμιση μόνο ικανοποιητική αυτή η διαπίστωση. Γιατί, διότι οι ανησυχίες που είχαν εκδηλωθεί μετά το κλείσιμο της ε, οδού των Δυτικών Βαλκανίων πως θα μετακινούνταν αυτές οι ροές προς τη Δυτική Μεσόγειο μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Βέβαια, στη Λιβύη αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αξιόπιστους συνομιλητές για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε στο βαθμό του δυνατού τα προβλήματα τα σχετικά με τους ε, πρόσφυγες. Αλλά υπάρχουν αντίστοιχε συνομιλίες με την Αίγυπτο και θα ήθελα ιδιαίτερα να επισημάνω προειδοποιητικά ότι θα ήταν φαινάκι να περιμένουμε ότι θα γίνουν ε, τα πάντα χάρη στο χρήμα, ότι μπορούμε να τα λύσουμε όλα. Δεν είναι δυνατόν ε, η εντύπωση να είναι πως η πλούσια Ευρώπη αγοράζει, εξαγοράζει τους φίλους της ανά τον κόσμο. Εμεί θέλουμε εταίρους, δεν θέλουμε ε, κάτι το οποίο αγοράζει το χρήμα. και γι' αυτό ε, μια πρωτοβουλία που θα αποτελούσε μια ε, εναλλακτική ε, σε σχέση με το, μια διαφορετική εκδοχή του σχεδίου Juncker και θα αφορούσε τέτοιες χώρες ώστε να συγκρατήσει τις μεταναστευτικές ροές σαν τελικό αποτέλεσμα θα ήταν ένας δρόμος, μία λύση αλλά μόνο εάν μπορέσουμε να πείσουμε τους ανθρώπους αυτούς, γιατί δεν μπορούμε να τους πείσουμε εξαγοράζοντας τους με χρήματα, αν μπορέσουμε να πείσουμε τους ανθρώπους αυτούς ότι έχουν επαρκείς οικονομικές συνθήκες ε, διαβίωσης εκεί, ώστε να μην χρειάζεται να εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους. Πράγμα το οποίο θα αποτελεί, βέβαια μεγάλη πρόκληση δεδομένων και των δημογραφικών εξελίξεων στην Αφρική, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε. Και βεβαίως πολύ μεγάλη σημασία έχει η πολιτική σταθερότητα στη Βόρεια Αφρική, πάνω στην οποία πρέπει να κάνουμε πολύ σοβαρή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο, κύριε Επίτροπε. Μια πρόταση για το δημοψήφισμα στη Ρεπούμπλικα Σέρψικα. Ε, ξέρουμε πολύ καλά πόσο καλή είναι στο να προετοιμάζουν εκλογές που τελικά δεν διεξάγονται. Ε, ας πούμε και ότι και αυτό το δημοψήφισμα μπορεί να το προετοιμάσουν, αλλά δεν θα το πραγματοποιήσουν εν τέλει. Σας ευχαριστώ θερμά για τη δεξιοδική αυτή παρουσίαση και συζήτηση. Και επισημαίνω ότι την προσεχή πέμπτη στις 8 έχουμε συνεδρίαση της Επιτροπής. Και όμως κύριε Γκάλερ, όντως, όντως, 8 η ώρα. Και με χαρά θα σας ξαναδώ. Με πρωινό μαζί, εντάξει. Να το οργανώσουμε. Όπως εκεί κυλαγκάρσα 1,5 ε, ε, μέτρο ύψος από το, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, Γεωργική Επιτροπή, που οργάνωνε πρωινά τέτοια με συναντήσεις με μπριζόλες, μπλάντι μέρη και ε, οχτώ τουλάχιστον ε, πιάτα. Μετά βέβαια το απαγορέψαν αυτό. Αλλά εμένα μου είχε δύο φορές να με παρόν εκεί. Ε, πρόγευμα εργασία το λέγανε. Σας ευχαριστώ.